Λεγκούτκο. Περνάμε στις ε, προτάσεις ε, ορισμού μελών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν έχει υποβληθεί καμία τροποποίηση, καμία αλλαγή. Συνεπώς ε, θεωρώ εγκεκριμένες τις προτάσεις της διάσκεψης των Πρόεδρων. Κύριε Χάρμς, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εχθές ε, μας ήρθε μια πολύ δυσάρεση είδηση, συγκεκριμένα από τον Κρόσνη, από την Τσετσενία. Συγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος, ε, η Ναστάλια Ισχυμίροβα, που είναι πολύ γνωστή σε εμά, δολοφονήθηκε. Τη βρήκαν νεκρή, αφού την είχαν απαγάγει πρώτα στον Κρόσνη. Τη βρήκαν λοιπόν νεκρή, λίγο μετά τα σύνορα ανάμεσα στην Τσετσενία και την Ιγκουσετία. Η Νατάλια Ζιαμίροβα εργάστηκε σκληρά στην Τσετσενία και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να ικανοποιήσετε το αίτημά μας που είναι να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τώρα για αυτή την ιδιαίτερα μαχητική δημοσιογράφο αμήντορα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία. Μάλιστα, κυρία Χάρμς.